όπως αναφέρεται στο άρθρο 211. Σε σχέση λοιπόν με τα κείμενα αυτά, βάσει του άρθρου 216 παράγραφος 4 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θεωρείται ότι γίνεται δεκτή η πληροφόρηση για τα θέματα αυτά, αν δεν υπάρξει μια αντίρρηση από πολιτική ομάδα ή 40 τουλάχιστον βουλευτές. Οπότε θα πρέπει να ψηφιστούν τα κείμενα αυτά. Τα κείμενα αυτά βρίσκονται στην ιστοσελίδα Seance on και αυτά θα καταγραφούν και στα πρακτικά της τέχουσα συνόδου. Ερχόμαστε τώρα στην για διάταξη, η οποία έχει αποφασίσει